θέση του στην πρώτη ανάγνωση για την οδηγία σε σχέση με τα πακέτα ταξιδιών και τις σχετικές ρυθμίσεις και τον κανονισμό που ορίζει κανόνες για την ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ και την περιαγωγή. Όλα αυτά θα περιλαμβάνονται στα πρακτικά της συνόδου αυτής και σε τρεις μήνες έχει, μάλλον και το Κοινοβούλιο έχει τρεις μήνες για να υιοθετήσει τη θέση του. Η προθεσμία ξεκινά από αύριο.